Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχηθώ ευτυχές στο νέο έτος. Έχουμε το καθήκον όχι μόνο να θυμίσουμε αλλά και να προστατεύσουμε τους νικητές αυτού του βραβείου του Ζαχάροφ που είναι σύμβολο όλων όσων αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα